Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίστε. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι εγκρίνετε την μέσα διάταξη και σας προτείνω να προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε την ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα για τη συνεδρίαση που προβλέπεται σήμερα βέβαια και για τη συνεδρίαση που προβλέπεται αύριο το πρωί πάλι να τα δούμε όλα σήμερα εκτός του σημείου 7 που αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο Juncker, επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Αυτή η ανακοίνωση προβλέπεται για τις 11 Δεκεμβρίου, δηλαδή για την 5η 11 Δεκεμβρίου. Κατά τα λοιπά όμως, ε, προτείνω να εξετάσουμε όλα τα σημερινά και τα βρενά θέματα της σημερινής διάταξης σήμερα. Έτσι θα κερδίσουμε χρόνο, επειδή ο τριμερής διάλογος συνεχίζεται και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει πάλι να συναντηθούμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, Το πρώτο σκέλος της συνεδρίασής μας θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Γι' αυτό παρακαλώ όσους δεν περιλαμβάνονται στο κεκλεισμένο των θυρών να μας αφήσουν για λίγο προκειμένου να συζητήσουμε μεταξύ μας τα σημεία 4, 5 και 6. Les points 4 et 5. Συγχωρείτε λέει στα σημεία 4 και 5. Νόμιζα και, ότι και το 6 ήταν και κλεισμένο το τυράννο. 4, 5 και 6, όχι. Bien, ça y est, le mouvement a eu lieu. Εντάξει. Όπως γνωρίζετε,